Okay, colleagues, we move to the Πάμε σε επεξηγήσει ψήφου. Ξεκινάμε με την έκθεση Νάταλι Γκρίσπακ Μπέκ. Ο πρώτο ομιλητή είναι ο κύριο Ντέβα. Ένα λεπτό. Κύριος Ντέβα. Είναι εδώ ο κύριος Ντέβα. Αν επιθυμείτε να μιλήσετε κύριε Ντέβα, μπορείτε να έχετε να πάρετε το λόγο. Αν όχι, δεν είναι υποχρεωτικό. Κυρία Πρόεδρε, ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που μας κληροδότησε η νομική μας παράδοση στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι η Μάγνα Κάρτα. Ότι κανείς δηλαδή δεν θα πρέπει να δικάζεται και να συλλαμβάνεται χωρίς λόγο και δεν μπορεί να κρατείται στη φυλακή για μεγάλο χρονικό διάστημα άνευ και αιτίας. Αυτή η παράδοση που όλοι, ακόμα και ο μονάρχης, οφείλει να τηρήσει, ήταν μία από τις πιο σημαντικές, από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα του νομικού μας ε, συστήματος, το τεκμήριο της αθωότητας. Είσαι αθώος μέχρι να αποδειχθείς ένοχος. Εάν έχουμε μια διαφορετική δομή, τότε το κράτος γίνεται κυρίαρχος εταίρος και ο πολίτης είναι ο κυδεμονευόμενος αυτή τη σχέση. Αν όμως το κράτος πρέπει να αποδείξει ότι είσαι ένοχος, η πολιτεία, τότε σημαίνει ότι τα δικαιώματα του πολίτη πριτανεύουν. Ευχαριστούμε κύριε Ντεβά. Η κυρία Μορβάη. Ευχαριστώ για το τεκμήριο αθωότητας. Είναι μια πολύ σημαντική έκθεση αυτή, την υπερψήφισα. Γιατί το τεκμήριο αθωότητας είναι μια αρχή πολύ σημαντική για τους πολίτες, ούτως ώστε να υπερασπιστούν τον εαυτό τους απέναντι στις υπερβολές της εξουσίας. Ειδικά όταν έχουμε μία υπόθεση στο δικαστήριο, όταν έχουμε μία σύλληψη, η οποία μπορεί να γίνεται λόγω πολιτικών κινήτρων, όπως συμβαίνει αυτό στη Ρουμανία. Στη Ρουμανία, ας πούμε, συλλαμβάνουμε Ούγγρους στην ε, υπόθεση Ντινότε Ιστφαν Μπέκερ. Είναι πολύ σημαντικό σε αυτήν την περίπτωση το τεκμήριο της αθότητας. Το βάρος της απόδειξης το φέρουν οι αρχές, αυτές που να αποδείξουν με αποδεικτικά στοιχεία ότι υπάρχει ενοχή από πλευράς του πολίτη. Το να συλλαμβάνεις κάποιον ή το να τον κρατάς στη φυλακή Ευχαριστώ μόνο ένα λεπτό είχατε κυρία μου. Ένα λεπτό μόνο. Κύριος Πόσπισερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ υπερψήφισα αυτή την έκθεση. Στη χθεσινή συζήτηση εξήγησα γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ενιαία δικονομία για τις ποινικέ δίκες στην Ευρώπη, όπως έχουμε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Δεν πρόλαβα όμως να πω ότι είναι καλό ότι υπήρξαν οι αναγκαίες αλλαγές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διότι βελτιώνει κατά πολύ το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διορθώνει κάποιες ε, αδυναμίες του. Βεβαίως πρέπει να μην υπάρχουν εξαιρέσεις το ότι το βάρος της απόδειξης το φέρει η εισαγγελία, το κράτος, όχι ο κατηγορούμενος. Και δεν ξέρω γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήθελε να παραβιαστεί αυτή η θεμελιώδης αρχή. Επίσης, ε, ορισμένες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς είναι η ποινική διαδικασία. Ευχαριστώ κύριος Μαμίκινς το τεκμήριο αθότητας ε, είναι ιδιαίτερα σημαντική αρχή στην δικονομία. Είναι σαν μία από τις δέκα εντολές και αυτό ισχύει παντού στον κόσμο. Η ιδέα λοιπόν είναι πολύ καλή και πρέπει οπωσδήποτε πάντα να εφαρμόζεται. Γι' αυτό στήριξα τη σημερινή μας απόφαση στις ποινικέ ε, διαδικασίες δεν πρέπει να υπάρχει κανένας καταναγκασμός και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και πρέπει οπωσδήποτε το βάρος ε, της απόδειξης ε, της ενοχής ε, να το φέρει η εισαγγελία. Θεωρώ ότι όλα αυτά είναι απόλυτα αναγκαία για το κράτος δικαίου. Τονίζω λοιπόν ότι υπερψήφισα αυτή την έκθεση διότι θεωρώ ότι είναι απολύτως αναγκαίο για την περαιτέρω εξέλιξη του δικαίου μας. Και εγώ υπερψήφισα αυτή την έκθεση και χαίρομαι ιδιαίτερα που ε, πέρασε με μεγάλη πλειοψηφία γιατί η πρόταση αυτή είναι πολύ θετική και φυσικά ε, οι δημόσιες αρχές δεν πρέπει να δίνουν ε, ενημέρωση στα μέσα μαζική ενημέρωση, εάν αυτό θα είναι ει βάρο του κατηγορουμένου και δεν πρέπει να επιτρέπεται κανένα καταναγκασμός για να ληφθούν στοιχεία από του κατηγορούμένου. και πρέπει να υπάρχουν πολύ αυστηροί περιορισμοί στι περιπτώσει που είναι δυνατόν να προχωρήσει η δίκη χωρί την παρουσία του κατηγορουμένου. Όλα αυτά είναι απόλυτα αναγκαία για να έχουμε ένα σωστό και δίκαιο σύστημα ποινική δικαιοσύνη και η ποινική δικονομία να είναι διαφανή και όσο δυνατόν πιο σαφή. Όλα αυτά εξαρτώνται επίσης γιατί συσχετίζονται με τις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σεβασμού των δικαιωμάτων όλων συμπεριλαμβανομένων των κατηγορουμένων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Χάναν. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 800 χρόνια πριν ορίσαμε τη αρχή του Χάμπεας Κόρπους, ότι δεν μπορεί κανείς να κρατείται ή να συλλαμβάνεται χωρίς λόγο. Και τώρα ε, χάρη στη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιλικής ε, Δικαιοσύνης και του εντάλματος ε, συλλήψεως, του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Συλλήψεως, αυτό δεν ισχύει πλέον. Ξέρω για έναν άνθρωπο ο οποίος δύο χρόνια παρέμεινε στις φυλακές της Ελλάδας για ένα ποινικό αδίκημα για το οποίο απαλλάχθηκε μόλις μπήκε στο δικαστήριο, διότι ήταν σαφές ότι δεν ίσχυε, δεν υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία. Όταν κρατείται κανείς ε, χωρίς να έχει κατηγορηθεί για δύο χρόνια είναι εντελώς ε, εσφαλμένο. Άρα δείχνουμε ότι δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να τιμωρούμε. Άρα σε αυτή τον ε, πανηγυρισμό της Μάγνα Κάρτα, τον υπάρχουν τέτοια στοιχεία και πράξεις, είναι κάτι το επονίδιστο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Από την έγκριση της Magna ε, Carta Libertatum ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας και γι' αυτό εμείς έπρεπε να δεχτούμε την εγγύηση μιας δίκαιας δίκης και στα ποινικά δικαστήρια, αλλά αυτό αφορά και την όλη ποινική διαδικασία που ορίζει τη βάση μιας δίκαιας δίκης. Σε ορισμένες χώρες αυτές οι αρχές ίσχυσαν για αιώνες και είναι αδύνατον να αποδυναμώσουμε ορισμένα δικαιώματα και εγγύησεις που απορρέουν από τη Συνθήκη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Αυτή είναι η βάση μιας δίκαιας δίκης. Γι' αυτό και θα ψηφίσω κατά αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στην έκθεση Φόρτ Μέσα Ατομικής Προστασίας Μαμίκεν. Αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχουν ε, μέσα ατομικού εξοπλισμού. Υπάρχει μία μακρά ιστορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 89 και μετά και λαμβάνουμε υπόψη και τις τεχνικές εξελίξεις. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι θα πρέπει να ε, αναθεωρήσουμε την οδηγία επικαιροποιώντα την, γιατί έχει μεγάλη σημασία για την κοινή αγορά. Θεωρώ ότι ο ατομικός εξοπλισμός προστασίας έχει μεγάλη σημασία για τους πυροσβέστες, για τους στρατιώτες και ούτω καθεξής. Χρειάζονται διαφορετικοί κανόνες ως προς την ποιότητα και τη χρήση. Νομίζω ότι η έκθεση αυτή είναι εξαιρετική και θα ήθελα να τονίσω ότι υπερψήφισα την έκθεση για άλλη μια φορά. Ο κύριος ε, Κέλλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε, και εγώ υπερψήφισα την έκθεση αυτή της κυρίας Φόρτ, η οποία έκανε μεγάλη, κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για την εργασία αυτή. Χαίρομαι ότι τώρα θα υπάρχει ένας κανόνας και αποτίμηση συμμόρφωσης για όλα τα προϊόντα έτσι ώστε οι αρχές εποπτείες της αγοράς να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει και η χρήση της επίσημης γλώσσας της χώρας εισαγωγέα και μια γλώσσα η οποία είναι ευνόητη για τους καταναλωτές. Συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι θα πρέπει οι κατασκευαστές να δίνουν σαφείς και κατανοητές οδηγίες χρήσεως και να ελέγχουν τις προδιαγραφές προστασίας. Άρα αυτό που έχει σημασία είναι η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα για να την έχουμε την στη δυνατή προστασία των πολιτών μέσα στα πλαίσια της, ε, του, της, του εξοπλισμού προστασίας. Χάναν. αποχώρησε. Πόλτσακ. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο, Πρόεδρε. Τα μέσα ατομικής προστασίας ε, πρέπει να ακολουθούν τις εξελίξεις τις τεχνικές. Υπάρχουν ε, και ευκαιρίες πέρα τους κινδύνους. Αυτά συνδέονται με τις αρχές της εσωτερικής αγοράς. Η βελτίωση των κανόνων για την ατομική προστασία θα επηρεάσει τον προϋπολογισμό των νομικών προσώπων, νομικών οντοτήτων, καθώς και των ατόμων που δουλεύουν για αυτές. Υποστήριξα αυτή την πρόταση και θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια για τη θαυμάσια δουλειά της. Αποφάσισα να συγκρίνω τα υπέρ και τα κατά τα οποία σας ανέφερα. Σε ό,τι αφορά την ε, προσωπική προστασία δεν πρέπει να χάσουμε την ευκαιρία που μας δίνουν οι νέες νομικές διατάξεις. Παρά λοιπόν κάποια προβλήματα που υπάρχουν, πιστεύω ότι θα πρέπει να κρατήσουμε ψηλά τα πρότυπα και να υποστηρίξουμε αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ. Πάμε στην έκθεση Στήλε, συσκευές αερίου, ο κύριος Μάμικενς. Κύριε Πρόεδρε, Πολλοί κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιούν ξύλο, πετρέλαιο ή βιολογικά απόβλητα για να θερμάνουν το σπίτι τους. Τα συστήματα που χρησιμοποιούν αέριο, που καίνε αέριο, είναι τα πιο δημοφιλή. Συχνά οι χρήστες βρίσκονται κοντά σε αυτές τις συσκευέ αερίου. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να βελτιωθεί η ασφάλεια των συσκευών αυτών. Γιατί μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει προβλήματα στην υγεία του από τις συσκευές αυτές, εάν δεν έχουν καλή συντήρηση. Η ενοποίηση και η τυποποίηση λοιπόν για τη χρήση αυτών των συσκευών στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια θαυμάσια πρόταση. Κύριο Ευχαριστώ. Όπως και με την προηγούμενη έκθεση, η συγγήτρια η Κάθριν Στίλερ πρέπει να επενεθεί για την έκθεση της αυτή ή την υπερψήφισα. Είναι σημαντική γιατί αλλάζουν κάποια πράγματα και ολοκληρώνεται έτσι η ενιαία αγορά ακούσαμε σήμερα το πρωί και από την Ολλανδική Προεδρία για το θέμα αυτό και είναι πολύ σημαντικό. Σε σχέση με το αέριο είναι πολύ σημαντικό, γιατί το αέριο θα είναι πολύ σημαντικό τμήμα, καθώς ακόμα και όταν περάσουμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ακόμα και τότε θα είναι σημαντικό το αέριο στο ενεργειακό μείγμα. Οι συσκευές αερίου πρέπει να σέβονται υψηλά πρότυπα γιατί μερικέ φορές ε, οι συσκευέ αυτές εκλείουν μονοξίδιο του άνθρακα που μπορεί να σκοτώσει. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να έχουμε την υψηλότερη δυνατή προστασία για τους καταναλωτέ. στις συσκευές αυτές. Η επόμενη ε, έκθεση είναι η εγκαταστάση με σειρματόσχηνα ε, Λόπες Ιστούρης White. Κυρία Άντερσον, η πρώτη ομιλήτρια. Υπάρχουν πολλές χιλιάδες ε, οχήματα τα οποία βασίζονται σε σηματόσχηνα και πρέπει να είναι ασφαλή και το κοινό να έχει κάθε εμπιστοσύνη στην ασφαλεία τους. Ο νέος κανονισμός αυτός θα ενισχύσει τις προδιαγραφές για την κατασκευή και το σχεδιασμό τους ιδιαίτερα σε αθλητικές εγκαταστάσεις και σε αστικές περιοχές. Ως υπεύθυνη για το θέμα αυτό από πλευρά τη πολιτική μου ομάδα, καλωσορίζω αυτέ τι ρυθμίσει και το γεγονό ότι ενεκρίθησαν με βρία πλειοψηφία και όλη την εργασία που έχει γίνει για να υπάρξει αυτή η βελτίωση του κανονισμού για τι εγκαταστάσει σύρματο χήνων, για να υπάρχουν σαφή κριτήρια και ισχυρότερε και βαρύτερε κυρώσει για να αντιμετωπιστούν παραβιάσει. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Παμίκινς. Κυρία Πρόεδρε. η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρωτοπορία σε αυτές τις εγκαταστάσεις σύρματοσχήνων και τη χρήση τους. Γύρω στις 1.700 εγκαταστάσεις ε, λειτουργούν στην Ένωσή μας που είναι το 60% της παγκόσμιας χρήσης και είμαστε και πρωτοπορία στην παραγωγή αυτών των ε, μηχανισμών και εξοπλισμών. Άρα είναι απόλυτα σκόπιμο αυτός ο νέος κανονισμός να βελτιώσει την υπάρχουσα κατάσταση. Νέες προδιαγραφές λοιπόν θα εφαρμοστούν και οι αναγκαίες τεχνικές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν. Αυτό είναι σημαντικό. Και είναι επίσης σημαντικό εγκαταστάσεις που έχουν και μια ιστορική αξία να μην θυγούν από αυτούς τους νέους κανόνες με τρόπο υπερβολικό. Γι' αυτό και υπερψήφισα και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κέλλη. Σας ευχαριστώ και πάλι κύριε Πρόεδρε, όπως και για τις προηγούμενες δύο εκθέσεις. Η έκθεση αυτή μας δίνει την δυνατότητα να εφαρμόσουμε και για αυτό το κλάδο την ενιαία ώρα και φυσικά την υπερψήφισα. Ήμουν παρόν χθε κατά την συζήτηση και πολλοί συνάδελφοι ε, εξέφρασαν την υποστήριξή τους προς αυτό το νομοθέτημα δεν είναι ίσως το πιο προβεβλημένο νομοθέτημα, δεν θα γραφούν πολλά άρθρα για τον εισηγητή, αλλά παρόλα αυτά βοηθάει ε, να αυξηθεί η ασφάλεια των πολιτών μας. Η εναρμόνιση των κριτηρίων για την ε, ασφαλή εγκατάσταση των ε, εγκαταστάσεων αυτών και την αγορά των συστατικών τους θα βοηθήσει και τους εργαζόμενους και τους πολίτες. Είναι καλύτερο επίσης να εξαιρεθούν οι ιστορικού τύπου εγκαταστάσεις από τον κανονισμό αυτό. Για άλλη μια φορά νομίζω ότι ο εισηγητής έκανε κάτι πολύ θετικό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χάναν ε, δεν είναι παρόν. Περνάμε στην επόμενη έκθεση η ειρνευτική διαδικασία στην Κολομβία. Ο κύριος Ποσπίσιν. Ευχαριστώ υπερψήφισα την πρόταση ψηφίσματος και θα ήθελα να λάβω το λόγο γιατί συχνά μιλάμε για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά τον κόσμο, μιλάμε για το πού και πότε υπάρχουν εμπόλεμες σειράξεις ή εμφύλοι πόλεμοι και εδώ έχουμε να κάνουμε με μία εξαίρεση. Καλωσορίζουμε μία ειρηνευτική διαδικασία στην Κολομβία με αυτή μας την πράξη. Γι' αυτό χαίρομαι που μπόρεσα να υπερψηφίσω αυτή την πρόταση γιατί μετά από 50 χρόνια εμφυλίου πολέμου σε αυτή τη χώρα της ε, Λατινικής Αμερικής υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ και η κυβέρνηση θα κάνει ανακοχή με τις άλλες εμπόλεμες ομάδες. Προετοιμάζαμε αυτό το κείμενο εδώ και τέσσερα χρόνια. Εάν εγκριθεί φέτος, τότε θα υπερισχύσει η ειρήνη στην Κολομβία. Μάμικενς. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι ο εμφύλιος πόλεμος στην Κολομβία ήταν από τους πιο μακροχρόνιους πολέμους στην σύγχρονη ιστορία. Εκατοντάδες, χιλιάδες θύματα ε, απομακρύνθηκαν από τις οικογένειές τους και ούτω καθεξής. Πέρσι συναντήθηκα με τον πρόεδρο της Κολομβίας ως μέλος της ε, αντιπροσωπείας από το ΕΛΚ και λάβαμε υπόψη το άρθρο υπαριθμών 5 της Γενικής Συμφωνίας. Αυτό είναι ένα πολύ καλό βήμα προς τα εμπρός. Αντιμετωπίσαμε πολλές δυσχέρειες Και αυτό αφορά και τις αντίπαλες ε, ομάδες. Υπήρχαν ε, διαπραγματευτές από την Χιλή, την Ορβηγία και την Αργεντινή. Ευτυχώς εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάναμε ένα βήμα προς το προς. Ο κύριος Χάνεν είναι απόν, άρα λίγη και αυτή η συνεδρίαση μέχρι τις 3 το απόγευμα. Αναστέλτε μέχρι τις 3 το απόγευμα. Σας ευχαριστώ πολύ.